δεν μπορεί να θεωρούν ότι μετά από την έγκριση συνθήκης Λισαβόνας δεν μπορεί να, μπορεί να αντιμετωπίζουν στο Κοινοβούλιο. Θυμηθείτε το SWIFT. Ευχαριστώ. Έχει κλείσει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη Σύνοδο Ολομέλειας στις Βρυξέλλες. Και τώρα. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι η έκθεση Simpson κοινοτικοί προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου. Μη εδώ του κυρίου Σίμψον θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Ελ Χαδράουι, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του εισηγητού για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Σίμψον, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα και γι' αυτό μου ζήτησε να διαβάσω τη δήλωσή του η αναδιατύπωση για την ανάπτυξη των προσανατολισμών ε, για, τα, για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών προσπαθεί να συνδυάσει ε, τις ε, διάφορες τροπολογίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και να ενσωματώσει και τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τη διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε 27 κράτη-μέλη. Οι προσανατολισμοί αναφέρονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Στόχο είναι μέχρι το 2020 να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο που να ενσωματώνει ε, τα δίκτυα υποδομή ε, αερομεταφορών, ε, θαλασσίων μεταφορών και μεταφορών στη ξηρά. Επειδή η Κομισιόν έχει κάνει κάποιες τροποποιήσεις στο παράρτημα ε, έπρεπε να εφαρμοστεί η διαδικασία τη αναδιατύπωση. Οι τροποποιήσει ε, στο παράρτημα έγιναν για να διορθωθούν κάποια ε, λάθη που έγιναν όταν προσχώρησαν τα νέα το 2004. Οι τροποποίησει δεν έχουν να κάνουν με την επικαιροποίηση των χαρτών, ούτε είναι τροποποιήσει επί τη ουσία. Οι δύο τροπολογίες του εισηγητή αναφέρονται σε κάποιε μικρέ αλλαγέ στα, στα εκτιμώντας. Πρόκειται γενικά για μικρέ μικρέ ε, τροποποιήσει ε, και έχουν να κάνουν με τη διόρθωση των ε, κατευθυντηρίων γραμμών. Ακολουθήσαμε τη Συμβουλή τη επιτροπή και δεν κάναμε αλλαγέ αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές. Σε αυτό συμφώνησε και η Επιτροπή. Ωστόσο, ο εισηγητή γνωρίζει ότι οι πράσινοι έχουν υποβάλει ε, μια τροπολογία που έχει να κάνει με την ε, ε, σύνδεση της πόλης του Μονάχου με το αεροδρόμιο. Αλλά θέλουμε να διορθώσουμε το κείμενο, όχι να το επικαιροποιήσουμε. Στόχος της αναδιατύπωσης είναι να μπουν όλα σε τάξη πριν την ε, ολική αναθεώρηση το 2011. Είναι, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη σαφήνεια των κατευθυντήριων γραμμών υπό το φως των πιο ουσιαστικών αλλαγών που θα γίνουν του χρόνου. Όλοι περιμένουμε την πραγματική αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών και τις ε, τάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων. Για να φτάσουμε εκεί όμως θα πρέπει να διορθώσουμε την παρούσα ε, νομοθεσία και ακριβώς αυτό κάναμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν έχει το λόγο, ο Επίτροπος Πίπαλης. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, τα λόγια του εισηγητού. Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Γι' αυτό δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Γιατί νομίζω ότι ο εισηγητής έχει περιγράψει επακριβώς τα διακυβευόμενα. Απλώς πω να σας πω πού βρισκόμαστε σε σχέση με την αναδιατύπωση, την αναθεώρηση, επί τη βάση Τη πράσινη Βίβλου το 2009, η Κομισιόν ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση με πάνω από 300 απαντήσει που λάβαμε και δημιούργησε έξι ομάδε εμπειρογνωμόνων για να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα τη διαβούλευση και να επεξεργαστούν μια νέα πρόταση πολιτική. Σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα λοιπόν θα υπάρξει μια πρόταση προς το Σώμα των Επιτρόπων το οποίο θα καθορίζει τη μεθοδολογία για το νέο διευρωπαϊκό δίκτυο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα μπορούσε να παρουσιαστεί στις 5 Μαΐου στο Σώμα των Επιτρόπων και μετά θα παρουσιαστεί προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η Κομισιό λοιπόν θα προχωρήσει προς την εκπόνηση προτάσεων για το νέο διευρωπαϊκό τι δίκτυο και τη χρηματοδότησή του. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτήν την ε, απόφαση από την πλευρά της Κομισιόν το πρώτο εξάμεινο του 2011. Ελπίζω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο κατανοεί την ανάγκη αυτών των αλλαγών και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή ε, συζήτηση σε σχέση με την αναθεωρημένη πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων με το Κοινοβούλιο του επερχόμενου μήνε. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε στου ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων από το ΕΛΚ, ο κύριο Σιλβέστρο, για δύο λεπτά. Ναι κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπε, εκφράζω ευγνωμοσύνη προς τους συναδέλφους που ακούγοντας τις προτάσεις και των σχεδόν συγητών και των συγητού ε, βοήθησαν να λήξει γρήγορα αυτή η υπόθεση και υπευλήθησαν τροπολογίες αν ήταν πάρα πολλέ όμω θα ήταν εμπόδιο για την υιοθέτηση αυτού του κειμένου κωδικοποίησεω. Είμαστε τώρα σε θέση να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη βάση για τον προγραμματισμό των διευρωπαϊκών δικτύων τη επόμενη δεκαετία για να είμαστε και πιο σύντομοι από την αρχή αυτού του θέματος κατέληξαν σε συμφωνίε οι ηγητέ να μην ε, υποβάλλουν τροπολογίε αν δεν έχουν συμφωνήσει το Συμβούλιο. Η Επιτροπή Μεταφορών έκανε τροποποίηση ε, τεχνική φύσεω κατόπιν επαφή με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και της, ε, του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι σε πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε να συμφωνήσει. Και συμφωνούμε με αυτή τη γραμμή που ακολουθήθηκε. Οι λίγε τροποποίησει που εκφράστηκαν επί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχουν αυτό το σκοπό και πιστεύω ότι είναι σκόπιμο για να έχουμε τελικό κείμενο που θα είναι συνεκτικό και σωστό. Ε, υποστημίζω γι' αυτό τις προτινόμενες τροπολογίες ενώ δεν θεωρώ ότι είναι έγκαιρη και σωστή η τροπολογία των πρασίνων που ήδη απερίφθη στη ψηφοφορία της στην Επιτροπή Μεταφορών. Η τροπολογία βρίσκει υποστήριξη όσον αφορά το περιεχόμενο, ατροποποιεί το χάρτη όσον αφορά το αεροδρόμιο του Μονάχου, και θα μπορούμε όμως να το δεχτούμε όταν μπούμε στι ουσίες αναλύσεως των διευρωπαϊκών δικτύων. Διότι οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τελικά θα προχωρήσουν γρήγορα. Αυτά σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές η κυρία Τικάο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Αυτό το έγγραφο επιτρέπει να επικαιροποιήσουμε το παράτημα 1 και το οποίο θα περιλαμβάνει τους χάρτες όλων των κρατών μελών, τους αναθεωρημένους χάρτες και προβλέπεται το 2020 ως ορίζον χρηματοδότησης όλων των σχεδίων. Για εφέτος προτείν, προτείνεται να υπάρχει ο χάρτης για όλα τα σχέδια TENT που περιλαμβάνουν τη Μαύρη Θάλασσα, την ε, Ουκρανία κτλ. ώστε να μπορέσει το δίκτυο υψηλής ταχύτητος να φτάσει στο Βουκουρέστι και στην Κωνσταντσα. Έχουμε δει ότι υπάρχουν σημεία τροτά στα συστήματα μεταφορών μας. Θα πρέπει να έχουμε τρόπους να μεταφέρουμε τους επιβάτες και σε άλλες μορφές διακίνησης όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα όπως σε αεροπορικές γραμμές. Είναι απαραίτητο λοιπόν το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας να φτάσει σε όλες τις πρωτεύουσες και τις μεγάλες πόλεις των χωρών μας. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να συνδέσουμε αυτές τις ενέργειες με την, ε, τις θαλάσσιες μεταφορές και τις εσωτερικές υδάτινες οδούς. Για τους πράσινους η κυρία Λίχτεμπέργκερ για δύο λεπτά. Μέρση κυρία Πρόεδρε. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την ολομέλειά μας και πρέπει να την απασχολήσει και στο μέλλον. Εδώ έχουμε μια αναδιατύπωση της οδηγίας και ο κύριος ε, Σιλβέστρος και άλλοι έχουν αναφέρει την έκπληξή τους που έχουν υποβάλει σχετικές τροπολογίες οι πράσινοι. Οι τροπολογίες των πρασίνων για την αλλαγή του, του καταλόγου των διευρωπαϊκών δικτύων αλλά δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι αυτό το οποίο έχουμε ψηφίσει, έχουμε ζητήσει εμείς αφορά μια ειδική περίπτωση εκεί που το ίδιο το κράτος μέλος είπε ότι αυτό το τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων το τρένο αυτό του Μονάχου δεν έχει πια νόημα. Είναι το περίφημο υπτάμενο μεταξύ του, της πόλης του Μονάχου και της, ε, του αεροδρομίου του, του Μονάχου. Νομίζω ότι κόλλησα ένα από τα σαρδάμ του κυρίου Στόιμπερ εδώ πέρα. Για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια επεξεργασία αυτών των δικτύων με μεγάλη προσοχή πρέπει να σκεφτούμε πάνω απ' όλα ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Πρόκειται για μία μελέτη κάποιου Ολλανδού, νομίζω γνωρίζετε αυτά κύριε Επίτροπε, μπορώ να σας τα δώσω, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τη μελλοντική συζήτηση. Και λέει ότι το κόστος ενός μεγάλου σχεδίου, και εδώ μιλάμε για πολλά μεγάλα σχέδια, γενικά κατά 45% υποτιμάται υποτιμάται κατά 45% και πάντα υπερτιμάται και η χρησιμότητα τέτοιων σχεδίων. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον υπολογισμό του κόστους των διευρωπαϊκών δικτύων και γι' αυτό <clears throat> σας καλώ να λάβετε υπόψη ότι τα θέματα αυτά είναι και δική μας ευθύνη να τα μεταφέρουμε και να πληροφορούμε σωστά τους πολίτες μας. Για τους φιλελεύθερους ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για μένα τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι ένα σημαντικό μέτρο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις παραγωγικές δομές της Ευρώπης. Στο νότο, στο βορρά, στη δύση, στην ανατολή είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε τις ιδεονομικές γραμμές και να μην αφήνουν τύφλα σημεία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε προς τα ανατολικά με αυτές τις γραμμές προς τις ε, χώρες της Ασίας και υπάρχουν και πολλές χώρες οι οποίες μπορούν με τον τρόπο αυτό να συνδεθούν με την Ευρώπη και να έχουν εμπορικούς δεσμούς. Η δημιουργία λοιπόν των, ευρωπαϊκών, διευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να στρέφονται και προς τα ανατολικά. Παραγωγός χάρη η σιδηροδρομική γραμμή η οποία περνάει από το Τσίσινάου και υπάρχει <clears throat> πρόταση να συνδεθεί <clears throat> έτσι η γραμμή Ουκρανίας στη Σνάου με την Βιέννη και με τις άλλες ευρωπαϊκές γραμμές, αυτό είναι κάτι το θετικό, το πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ κύριε Σόπερμαϊερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, προτιμώ να λέτε ότι είμαι χωρίς πολιτική ομάδα ε, από τη μία εγγεγραμμένος ελεύθερος από πολιτική ομάδα. Ε, έχουμε τώρα την ε, ευκαιρία να αναφερθούμε σε ε, ένα ιδιαίτερα προβληματικό έργο για την Αυστρία. Έχουμε το τούνελ και την σύνδεση Βερολίνου-Παλέρμο και τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το οποίο θα περάσει από τον άξονα Ινσπρουχ-Πότσεν η Αυστρία, το Τιρόλο, η Βόρεια Ιταλία και η Νότια Γερμανία εξαρτώνται από αυτό και ε, υπάρχει ο κίνδυνος ε, να δαπανηθούν ε, δισεκατομμύρια. Αρχικά το 2002 υπολογίζαμε δαπάνες δισεκατομμυρίων αλλά έχει εκραγεί το κόστος και τώρα μιλάμε για 16 δισεκατομμύρια. Η χρηματοδότηση δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα και το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τα εμπλεκόμενα εμπλεκόμενα εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα μετά το 2013, έτσι ε, τα, σχετικά, τα εμπλεκόμενα απλά περιμένουν. Και ε, θα πρέπει να εξεταστούν και οι δρόμοι προσέγγισης και η χρηματοδότηση και από ιταλικής πλευράς δεν, είναι, δεν έχει ξεκαθαριστεί η έκκλησή μου είναι λοιπόν ε, τώρα, εάν ε, προγραμματίσουμε τα δίκτυα ε, δεν μπορούμε να κάνουμε ανεπαρκή προγραμματισμό. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει με το 15% και θα πρέπει να προωθήσει το έργο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στους άλλους ομιλητές. Ο κύριος Κούν για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, οι προσανατολισμοί για την ανάπτυξη των ε, ε, διευρωπαϊκών δικτύων ε, είναι ένα θέμα που ακούγεται πολύ τεχνικό. Ο εισηγητής, ο κύριος Σίμψον, είπε ότι είναι ουσιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη στο μέλλον. Οι δρόμοι μεταφορών είναι οι φλέβες της οικονομίας και θα πρέπει να φροντίσουμε η Ευρώπη ως οικονομικός χώρος να μπορεί να συγκριθεί με ανάλογους ε, χώρους ε, ε, στι Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ασία. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις εσωτερικές μεταφορές, με ναι, να συνδέσουμε την Ευρώπη με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και να τα ενισχύσουμε. Οι μεταφορικές αρτηρίες στόχο έχουν να ε, μεταφέρουν τα προϊόντα εκεί που βρίσκονται οι πελάτες και Σημαντική είναι η ανάπτυξη ε, σημαντικών ε, μεταφορικών αρτοριών ώστε να προωθηθεί η οικονομία και δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Η Ευρώπη είναι ήπειρος με πολλές ακτές, με πολλά λιμάνια. Θα πρέπει να συνδέσουμε μεταξύ τους τα λιμάνια και θα πρέπει να, μην ξεχνάμε ότι η κινητικότητα είναι το α και το ω. Θα, πρέπει όμως να σκεφτούμε ε, και... Ε, το περιβάλλον. Αυτό στο μέλλον θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Ε, αποφασιστικής ε, σημασίας ερώτημα είναι μπορούμε να τι ε, συνδέσει Βορρά, Νότου και Ανατολή ε, Δύση που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορούμε να ε, τι μετατρέψουμε σε ένα δίκτυο. Διότι θα πρέπει να σκεφτούμε όταν δούμε τον, την βασική αρτηρία Παλέρμο-Βερολίνο μπορούμε να την επεκτείνουμε περαιτέρω ώστε να φτάσει στη Σκανδιναβία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιάλα Σέντερ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας είναι μια εδραίωση και της διαδικασίας εφαρμογής των διευρωπαϊκών δικτύων που θα μας προετοιμάσουν για την προηγούμενη, για την προτελευταία και τελευταία ε, μεταρρύθμιση ενώπιση του 2020 για να έχουμε μια καινοτόμα κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε ήδη συζητήσει για το θέμα του εκτελεστικού φορέα, έχουμε την άποψη όλων των συντονιστών και ελπίζουμε ότι θα συμπληρωθούν όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα θέματα που θέλουμε. Υπάρχει μεγάλη προστοκία από τους γείτονές μας, ιδίως στη Μεσόγειο, σε σχέση με αυτές τις πρωτοβουλίες για τα δίκτυα αυτά. Ελπίζουμε και αδειμονούμε αναμένοντας την πρόταση της Κομισιόν για τη μεθοδολογία η οποία θα μπορέσει να συμπληρώσει τη διαβούλευση και τη συζήτηση που κάναμε πρωτού προχωρήσουμε σε, μια, σε από τα πιο συναρπαστικά εγχείρηματα. Είναι απαραίτητο να έχουμε ένα δίκτυο κινητικότητας και συνοχής που θα εξασφαλίσει δυναμικότητα και είναι ο χώρο μεταφορών στην Ευρώπη των 27 εντοπίζοντας τα αεροδρόμια και τους κόμβους στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνοντας ως τα σύνορα και εξασφαλίζοντας την οσμοποίηση και την αλληλοδιαπερατότητα όλων των μορφών μεταφοράς και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να δημορφώσουμε ένα σχέδιο για την Ευρώπη του 2020 του 21ου αιώνα που θα έχει την απαραίτητη ακτινοβολία και χρηματοδότηση. Αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε ενώπιον μας. Προς το παρόν εμείς πρέπει να εγκρίνουμε αυτή την πρώτη νομοθετική πρόταση και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο μας τον κύριο Σίμψον για την πρότασή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κράμερ για να μισή λεπτό επίσης. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, το Transrapid δεν υπάρχει μέσα σε αυτήν την οδηγία. Δεν υπάρχει πια στο τοπίο. Δεν ε, έχουμε ενιαία συστήματα, έχουμε συστήματα τα οποία πολλαπλασιάζονται σε ποικιλία. Θα δοθούν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ποικίλα στέχεια, σχέδια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πει όχι στο Transrapid. Αλλά αναφέρθηκε και πάλι το 2006 σαν σχέδιο μεταφοράς μεταξύ Βερολίνου και, Αμβούργου. Το 1996 μετά εμφανίζεται σαν μια λύση μεταφοράς μεταξύ του αεροδρομίου του Μονάχου και του κυρίου σιδηροδρομικού σταθμού του, του... του Μονάχου. Κανείς δεν το θέλει λοιπόν, ούτε καν η βαβαρική κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργό τη ε, Βαβαρία, ο Έντμουν Στόιμπερ, προσπάθησε μετά από την έξοδό του από την κυβέρνηση της να αγωνιστεί για την κατάλυση τη γραφειοκρατίας στην Ευρώπη. Αλλά είναι δική του ευθύνη. Αυτό θα πρέπει μέσα στα πλαίσια αυτά να καταλάβει ότι δεν έχει καμία θέση το Transrapid στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα πρέπει να βγει. Ήταν πολύ καλό επιστημονικό παιχνίδι, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με την Ευρώπη είναι ένα ξένο σώμα και τα ξένα σώματα δεν έχουν καμιά σχέση σε αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάχτφιντ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Σίμψον και να εκφράσω την ε, λύπη μου που δεν μπορεί να είναι εδώ παρόν σήμερα. Ε, αλλά παρόλα αυτά συζητάμε το θέμα θα ήθελα να τον συγχαρώ για τη θέση του να αφήσει λίγο πολύ τα πράγματα όπως είναι ε, όσον αφορά την οδηγία αυτή. Ένα ε, θέμα είναι σημαντικό η αξιοπιστία για τον, Ευρωπαϊκό νομοθέτη, Ευρωπαίο νομοθέτη και ε, αυτό πληρούνται εδώ. Μία δεύτερη παρατήρηση. μία έκκληση και για το μέλλον όταν θα, αποφασίσουμε, όταν θα λάβουμε αποφάσεις για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Κάποιοι ε, επιχειρηματολογούν ε, υπέρ κάποιων συνδέσεων, άλλοι είναι κατά, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ποια ε, προσθέμενη αξία επιφέρει και τι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Τι θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει τελικά, διότι όταν τελικά εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά θα υποφεληθούν οι Ευρωπαίοι, οι επιβάτες και τα κράτη-μέλη που δεσμεύονται ε, να μεταφέρουν τις ε, μεταφορές από τους δρόμους ε, στους σιδηροδρόμους. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε τους ομιλητές στη διαδικασία Catch the Eye. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Μούλσερ για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, με το άνοιγμα προς την Ανατολική Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση η Βαλτική κερδίζει σε σημασία ε, μιλάμε για τον άξονα Βαλτικής Αδριατικής ε, και ε, από το Γκτάνς και προς την Τσεχία έχει επιβεβαιωθεί η σημασία του άξονα αυτού. Τώρα μιλάμε για επέκταση μέχρι την Ιταλία και στο δίκτυο αυτό το οποίο μεταφέρει το μισό περίπου όλων των αγαθών και των ανθρώπων στον άξονα αυτό θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν. Όπως ε, όλοι γνωρίζουμε, με την ε, αύξηση των ε, μεταφορών αυξάνεται και η τιμή και μόνο με την επέκταση του νότιου αυτού διαδρόμου και μεταφορά των μεταφορών από τους δρόμους στους σιδηροδρόμους θα έχουμε κάποιο όφελος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπαζέσκου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δοθέντως ότι αυτή τη στιγμή όλες οι αεροπορικές ε, τα αεροπορικά δρομολόγια έχουν διακοπεί λόγω της εκρήξεως του ηφαιστείου στην Ισλανδία, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό ε, δίκτυο μεταφορών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τις υποδομές των μεταφορών. Οι διασυνδέσεις μέσω αυτών των υποδομών στους κύριους άξονες που υπάρχουν, τους μεταφορικούς στα κράτη-μέλη και κυρίως στα νέα κράτη-μέλη είναι κάτι σημαντικό. Στη Ρουμανία έχουμε τρεις διαδρόμους διευρωπαϊκούς, τον 4, 7 και 9 και φτάνουν μέχρι το λιμάνι της Κωνσταντζας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο διάδρομο υπαριθμών 7, διότι ο Δούναβης είναι πρωταρχικός άξονας του δικτύου αυτού. Συνδέει τη Βόρεια Θάλασσα με τον Εύξηνο πόντο, το Ρότερντα με την Κωνσταντζα και θα μπορούσε να γίνει σπονδυλική στήλη πραγματική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Όλα μου χρειαζόμαστε συνεργασία για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτού του διαδρόμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Μάισνερ. Κυρία Πρόεδρε, πράγματι τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, εξυπηρετούν τι γενικέ μεταφορέ στην Ευρώπη. Δεν μπορεί, κανείς να πει ότι οι οι μεταφορές ε, είναι η σπονδυλική στήλη τη εσωτερική αγορά που αποτελεί ένα από του βασικού μας στόχου τη Ευρώπη και γι' αυτό είναι απαραίτητο να προσέξουμε να υπάρχουν πράγματι όλοι οι διάδρομοι εκεί που υπάρχει οικονομική ανάγκη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί ακριβώς σε αυτούς. Και φυσικά υπάρχουν πάντα εθνικά συμφέροντα. Ήδη βλέπουμε ότι κάποιοι μιλάνε για το Δούναβι, κάποιοι μιλάνε για την ε, Νότια Ευρώπη, άλλοι μιλάνε για το, για, το τούνελ Μπρέν Βάζλ. Παντού υπάρχουν ε, οι άξονες αυτοί και ε, σημαντικό είναι να περνούν μέσα από όλη την Ευρώπη ώστε να μεταφέρουν όχι μόνο τα αγαθά αλλά και τους ανθρώπου. Ε, από το Α στο Β. Αυτό είναι το καθήκον μας. Ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις περιφερειακές ε, συνθήκες για κάτι τέτοιο. Και σημαντικό είναι να έχουμε ένα λειτουργικό δίκτυο για όλα τα μέσα μεταφοράς. Αυτό είναι το θέμα και ακριβώς αυτό θα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάφμαν είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναφέρθηκε το το πέρασμα του Μπρένερ και η νέα διαδρομή μεταξύ του Μονάχου και της Βερόνας υπάρχει μεγάλη μεταφορά εμπορευμάτων από αυτό τον διάβλο και επομένω είναι απαραίτητο να γίνει το ταχύτερο δυνατό και από τις δύο πλευρές και από την Αυστρία και από την Ιταλία να γίνει χρηματοδότηση η οποία είναι απαραίτητη για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Δυστυχώς είναι δύσκολη χρηματοδότηση και από τις δύο πλευρές είναι απαραίτητο να μεταφερθούν να υπάρξει χρηματοδότηση των μεταφορών από τον αυτοκινητόδρομο στο τρένο. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία θα διατηρήσει την αποκλειστική εκμετάλλευση για άλλα 50 χρόνια. Επομένως δεν υπάρχει αυτή η διασταυρούμενη χρηματοδότηση και δεν μπορεί να εκμεταλλευτούμε όλα τα πλεονεκτήματα αυτή τη διάλευση. Η κυρία Γιάλα Σένερ. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει αυτή την αναδιατύπωση τη οδηγία για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα ήθελα η Κομισιόν να μου απαντήσει ώστε να το πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα του πότε θα έχουμε πρόσβαση στην ε, ανακοίνωση τη Κομισιόν για τη μεθοδολογία. Όπω ξέρετε κύριε, κύριε Επίτροπε, αυτό είναι μια από τι προτεραιότητε τη Ισπανική Προεδρία. Περάσαμε τον Ισημερινό, έχουμε περάσει το σημαντικό ορόσημο και πρέπει να ξέρουμε πια πότε θα μπορούμε να έχουμε αυτή τη μεθοδολογία για την έκθεση αυτή για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ενόχημα της Κομισιόν. Πάλι ο κύριος Επίτροπος Πίμπαλξ έχει το λόγο, εξ Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξανά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Μεταφορών. Την ευχαριστώ για την υποστήριξή της, γιατί αυτήν τεχνική αναδιατύπωση και ελπίζω ότι στην Ολομέλεια θα υποστηρίχει το κείμενο. Η σημερινή συζήτηση ε, ήταν ευρύτερης κλίμακας και θα βοηθήσει να προτείνουμε μια μεθοδολογία. Ο συνάδελφος αντιπρόεδρος Κάλλα στις 5 Μαΐου θα στείλει το κείμενο στο Σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαστήκαμε κάποιο χρόνο η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καινούρια βλέπετε και χρειάζεται κάποιο χρόνο το νέο σώμα να ετοιμάζει πρότασεις. Πιστεύω όμως ότι αποκομίζω από τη συζήτηση ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ένθερμα τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τις σχετικές πολιτικές. Διότι αυτές οι υποδομές διασυνδέσεων και στις μεταφορές και στην ενέργεια και στις τηλεπικοινωνίες αυτά τα δίκτυα ε, χρειάζονται να μιλάμε για την Ευρώπη. Θα μας βοηθήσει λοιπόν αυτή η συζήτηση να αναπτύξουμε μεθοδολογία. Σημαίνει λοιπόν ότι η Επιτροπή Μεταφορών θα έχει την ευκαιρία να το συζητήσει αν όλα πάνε καλά τον Μάιο. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι ο κύριος Ελχαδραουή, ο οποίος αντικαταστά τον κύριο Σίμψον ο εισηγητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη συζήτηση και να επαναλάβω ότι θέλουμε να διορθώσουμε σφάλματα που έγιναν κατά το παρελθόν και όχι να επιφέρουμε ουσιαστικές αλλαγές. Αυτό θα ακολουθήσει αργότερα όταν θα γίνει πραγματική αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών και προσβλέπουμε σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό το λόγο ο εισηγητής ο κ. Σίμψον και ο υποφαινόμενος ως εισηγητής της ομάδας μου θα ε, πούμε στην πολιτική μας ομάδα καταψηφίσουν την τροπολογία που υπέβαλαν οι πράσινοι και ελπίζω και άλλες πολιτικές ομάδες να μας υποστηρίξουν επ' αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη Ολομέλεια στις Βρυξέλλες. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Φαντάλεν «Στρατηγική στόχη και συστάσεις πολιτικής για τις θαλάσσιες μεταφορές της